της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για την απόφαση της ε, Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας να άρει την ασυλία 138 βουλευτών. Ευθύς εξ αρχής θα ήθελα να σας πω το εξής. Έχουμε καθυστερήσει και οι περισσότεροι ομιλητές, διότι υπάρχει μακρύς κατάλογος ομιλητών, έχουν ένα λεπτό στη διάθεσή τους και θα ήθελα να σας ζητήσω να τηρήσετε αυτό το ένα λεπτό διότι σκοπεύω και εγώ να τηρήσω τους χρόνους με μεγάλη αυστηρότητα. Θα ήθελα λοιπόν τώρα να δώσω το λόγο στον Επίτροπο Χάν για να ξεκινήσουμε τη συζήτηση. Ο Επίτροπος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θα ήθελα καταρχάς να ευχαριστήσω, να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια για τα θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία. Και θα ήθελα να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη στήριξη που μας δίνει ε, σε αυτή τη συνεργασία, στην ατζέντα που έχουμε με την Τουρκία, όπως αναφέρεται στο σχετικό ψήφισμα του Απριλίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δείξει τη βούληση που έχει να δώσει νέα πνοή στις σχέσεις με την Τουρκία στεναρά προσιλωμένη Ευρωπαϊκή Ένωση στις αρχές και στα κριτήριά μας και πρέπει να είμαστε στο ύψος της πολιτικής δέσμευσης που έχουμε αναλάβει ε, για την προόδο σε όλους αυτούς τους τομείς. Έγιναν συνομιλίες για θέματα οικονομικής στήριξης, εμπορίου, ενέργειας, ε, για, τις, ε, για το μέσο επίλυσης και διαχείρισης της προσφυγικής κρίσης 250 εκατομμύρια έχουμε δεσμεύσει, άλλα τόσα βρίσκονται επιτάπητος και αυτό δίνει προοπτική στους πρόσφυγες και απαλύνονται οι μεταναστευτικές πιέσεις. Όλα αυτά λαμβάνουν χώρα με βάση τα σημεία αναφοράς τα οποία υπάρχουν από το 2013 και δεν έχουν αλλάξει. Δεν είναι ε, μίας κατεύθυνσης ο δρόμος αυτός, ε, δεν είναι μίας κατεύθυνσης η πορεία αυτή, βασίζεται σε ένα ανοιχτό επικοδομητικό διάλογο και θα πρέπει να ειδωθεί στο ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο συμπεριλαμβανομένων των πολύ σοβαρών εξελίξεων στην Συρία. Παραμένει βασικός εταίρος στη διαχείριση της μετανάστευσης η Τουρκία. Η Τουρκία έχει κάνει πολλά για να βοηθήσει τους πρόσφυγες που χρειάζονται καταφύγιο ε, τρόφιμα, ζήτηση και ε, υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, διάφορες εξελίξεις και μάλιστα σοβαρές επηρεάζουν ε, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου Τουρκία. Σε, για όλα αυτά τα θέματα στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2015 για την Τουρκία εμείς ανέκαθεν είχαμε υποστηρίξει μια ξεκάθαρη θέση και αυτό φαίνεται και με το δικό σας ψήφισμα εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τις σοβαρές της ε, ανησυχίες για την άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας των βουλευτών, πολλών βουλευτών ε, της ε, Εθνοσυνέλευσης. Έχω έρθει σε επαφή με την Αντιπρόεδρο κυρία Μογκερίνη και στις 20 Μαΐου ε, καταστήσαμε σαφές ότι η ασυλία πρέπει να ισχύει για τους πάντες σε, επί τη βάση μη διακρίσεων. Αυτή είναι η σταθερή και συνεπής και μόνιμη στάση και απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και κάθε απόφαση για την άρση ασυλίας θα πρέπει να λαμβάνεται με βάση την εκάστοτε περίπτωση και σύμφωνα με διαφανή κριτήρια και όχι πολιτικές επιδιώξεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανειλημμένως το έχει ε, επαναλάβει αυτό και το πλαίσιο για την κοινοβουλευτική ασυλία θα πρέπει να περιλαμβάνει πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για την άρση αυτής όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλα τα ευρωπαϊκά κοινοβούλια στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και με συστηματικό τρόπο έχουμε τονίσει ότι είναι προβληματική η ερμηνεία του νομικού πλαισίου ε, αντισυνταγματική που ε, παρακολεί ε, την ελευθερία έκφρασης των μελών του Κοινοβουλίου στην Τουρκία. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι θα πρέπει κάθε ισχυρισμό για δίκαιμα που να έχει τυχόν διαπράξει βουλευτής του Τουρκικού Κοινοβουλίου ε, θα πρέπει να εξετάζεται αυτός ο ισχυρισμός σύμφωνα με τα κατάλληλα ε, κριτήρια, τα νομικά ε, κριτήρια διαφάνειας μεταξύ άλλων. Να τηρούνται τα δικαιώματα του ενδιαφερομένου αλλά να τηρούνται τα δικαιώματα και προς όφελος του ενδιαφερομένου και προς όφελος της σταθερότητας της χώρας. Η Τουρκία έχει ξεκινήσει μια πορεία προς την οικονομική πρόοδο. Ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε το θέμα στενά και θα θέσουμε αυτά τα ζητήματα στην επικείμενη συνάντηση υψηλού επίπεδου. Και καλούμε εν γέννη την τουρκική κυβέρνηση να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις σύμφωνα με τα δημοκρατικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ε, δουλεύουμε ε, γρήγορα ε, και με ταχύ ρυθμό για να έχουμε τα κατάλληλα προπαρασκευαστικά έγγραφα. Βεβαίως με την επιφύλαξη της θέσης των κρατών μελών σύμφωνα με τους υφιστάμενους Πιστεύουμε ότι ο ορισμό σημείων αναφορά στο δικαστικό πεδίο και στο πεδίο των θεμελιωδών δικαιωμάτων, των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τη ασφάλεια, τη ελευθερία, τη δικαιοσύνη. Αυτό είναι ο κατάλληλο τρόπο για να πείσουμε την Τουρκία να έχει ευρωπαϊκή προοπτική, να προσερκίσει την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και καλό ε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να στηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτό το εγχείρημα. Σα ευχαριστώ. Σα ευχαριστούμε, Επίτροπε. Θα ήθελα τώρα να ζητήσω να παρέμβει ο κύριος Πρέντα. Ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η άρση της ασυλίας ενός βουλευτή δεν είναι κάτι το εξαιρετικό για ένα κοινοβούλιο. Κάθε κοινοβούλιο το κάνει και εμείς το κάνουμε ε, στο Στρασβούργο. Όμως να αέρουμε την ασυλία 138 βουλευτών ταυτοχρόνως, ε, αυτό είναι έξω από τα συνηθισμένα. Και μάλιστα αποτελεί ένα εξαιρετικό γεγονός, πόσο μάλλον αφού οι βουλευτές αυτοί είναι όλοι από το κόμμα της αντιπολίτευσης, το κουρδικό, ε, που είναι αντιπολίτευση στην στην Επομένως υπάρχει αμφιβολία η οποία οφείλεται λόγω του συλλογικού χαρακτήρα της απόφασης αυτής και λόγω του αντίκτυπου που θα έχει αυτή η απόφαση στην εκπροσώπηση των πολιτών κουρδικής καταγωγής. Ε, σίγουρα έχουμε εταιρική σχέση με την Τουρκία για τους μετανάστες, για τις ε, θεωρήσεις, για τη διαπραγμάτευση, για την ε, προενταξιακή της πορεία. Όμως θα πρέπει να κρατήσει το λόγο της η Τουρκία για να σε σεβαστούμε και εμείς ε, τη δική μας ε, πλευρά της συμφωνίας. Ο κύριος Πύρη παρακαλώ. Η κυρία Πύρη, με συγχωρείτε. Σήμερα έγινε η, η τελετή των αστυνομικών που έχασαν, η κηδεία των αστυνομικών που έχασαν τη ζωή τους ε, χθε στην Κωνσταντινούπολη. Καταδικάζω όλες τις τρομοκρατικές επιθέσεις και εκφράζω τα θερμά μου και ειλικρινή συλληπιτήρια στα θύματα των επιθέσεων. Δεν μπορούν να υπάρξουν δικαιολογίε για τις φρικτές αυτές επιθέσεις. Θα πρέπει να γίνουν σωστές επενδύσεις και σωστά εγχειρήματα για να βρεθεί μία λύση στο κουρδικό και αυτό είναι προ όφελο της Τουρκίας και των πολιτών που κατοικούν στο νοτιοανατολικό άκρο της χώρας. Μας ενδιαφέρει ιδιαιτέρως η απόφαση άρσης ασυλίας του ενός τετάρτου των μελών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, πόσο μάλλον που ανήκουν όλοι αυτοί στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης ΧΑΝΤΕΠΕ πάρα πολλοί ε, κάτοικοι δεν μπορούν πλέον να εκπροσωπηθούν στην Εθνοσυνέλευση και δεν θεωρούμε ότι πρέπει να υπάρχει ασυλία ε, σε κάθε περίπτωση. Δεν θεωρούμε ότι δεν αντιμετωπίσει απειλές τρομοκρατικές η Τουρκία. Βεβαίως και ισχύουν όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά προσπαθούν να σιωπήσουν τους αντιπάλους λόγω των πολιτικών τους απόψεων και με αυτό δεν μπορούμε να είμαστε σύμφωνοι. Ε, θα υπάρχει σε δημοκρατικό εκλεγμένο κοινοβούλιο χώρος έτσι ώστε να γίνονται ανεκτές οι αντίθετες θέσεις. Όλοι έχουν κάνει λάθη. Είδαν, είδαμε φωτογραφίες ε, βουλευτών του ΧΑΜΤΕΠΕ να πηγαίνουν στην κηδεία ε, μελών ε, του ΠΚΚ. Πολλές φορές η εκεχηρία δεν έχει τηρηθεί. Έχουν γίνει λάθη από όλε τι πλευρές και υπάρχει απογοήτευση από όλε τι πλευρές. Αυτό είναι κατονοητό, αλλά πρέπει κανείς να κοιτάζει προ τα εμπρό Ένα εξόριστο κοινοβούλιο δεν μπορεί να είναι λύση. Ούτε μπορούν να είναι λύση οι στρατιωτικές παρεμβάσεις. Όλα αυτά έχουν αρνητικό αντίκτυπο στις ευρωτουρκικέ σχέσει και στις επόμενες εβδομάδες δημοκρατικώς ερετά εκλεγμένα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εξαφανίζονται πίσω από σίδερα, πίσω από κάγκελα με βάση μια, μια τρομοκρατική νομοθεσία εξαιρετικά αμφιλεγόμενη και αυτό θα παρακολουθεί θα παρακολύσει τη διαδικασία θεωρήσεων. Δεν μπορούμε να δεχθούμε δημοσιογράφοι πανεπιστημιακοί, μέλη του Κοινοβουλίου να ρίχνονται στη φυλακή γιατί έχουν εκφραστεί ελεύθερα. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συμβάλλει θετικά στην επανέναρξη της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία όμως οφείλει να ξεκινήσει στην ε, ε, Τουρκία καταρχάς. Και το λογικό είναι να ξεκινήσει από τη Βουλή, από την Εθνοσυνέλευση. Απευθύνω έκκληση σε όλες τις πολιτικές δυνάμεις της Τουρκίας από κοινού να κάνουν δήλωση κατά της τρομοκρατίας, να σταματήσουν την αιματοχυσία για χάρη όλων των πολιτών. Ευχαριστούμε ο κύριος Μαριάς για ένα λεπτό. Η συνεχίζει ακάθεκτα την πορεία του προς τον ολοκληρωτισμό, καθώς αποφάσισε άρση ασυλίας 138 δημοκρατικά εκλεγμένων εκπροσώπων του λαού, γιατί εκφράζουν τη φωνή 25 εκατομμυρίων Κούρδων που ζουν στην Τουρκία σαν να μην έφτανε αυτό οι τουρκικές αρχές αποφάσισαν να τελέσουν ισλαμική λειτουργία στην αγιά σοφιά προσβάλλοντας έτσι την πίστη εκατομμυρίων χριστιανών σε όλο τον κόσμο. κύριε χαν έχω ήδη αποστείλει στην κυρία μογκερίνη επιστολή με την οποία ζητώ την παρέμβασή της εδώ και τώρα για να σταματήσει αυτή η πρόκληση αυτή η βεβήλωση του ναού της ορθοδοξίας της αγιάς σοφιάς όπου κάθε μέρα γίνεται πλέον ανάγνωση του κορανίου. κύριε χαν η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει επιτέλους να πάψει να εθελοτυφλεί μπροστά στον αυταρχικό κατήφορο της τουρκίας μπροστά στις προκλήσεις της απέναντι στη χριστιανοσύνη. κύριε χαν ήρθε η ώρα η ευρωπαϊκή ένωση να πάψει να υποκλίνεται στο σουλτάνο. ευχαριστώ. Ο παρακαλώ στη συνέχεια. Ναι, σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Όλοι είμαστε κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, βουλευτές εδώ και φυσικά υπάρχουν καταστάσεις όπου η ασυλία ενός συναδέλφου πρέπει να αρθεί. Όμως η άποψη ότι εμείς ως κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να δεχθούμε την άρση ασυλίας εκατοντάδων βουλευτών λόγω λέει αδικημάτων ή παραπτωμάτων που ξεκινούν από μικρολεπτομέρειες μέχρι σοβαρότατες κατηγορίες, αυτό είναι κάτι το, το, το παρανοϊκό. Δεν είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι κάτι περισσότερο από εκπληκτικό ότι αποφάσισε η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση κάτι τέτοιο. Και είδα και τα κριτήρια της Κοπενχάγης ε, για την ε, Τουρκία, για μια χώρα που θέλει να γίνει κάποτε πλήρες μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο κριτήριο της, ε, των κριτηρίων της Κοπενχάγης σύμφωνα με το Eurolex είναι σταθερότητα θεσμική της, ε, του κράτους δικαίου, της δημοκρατίας, ε, προστασία μειονοτήτων. Αν ένα κοινοβούλιο το ίδιο αυτοκαταργείται και δεν είναι πλέον ε, ε, όργανο που να εκπροσωπεί τους πολίτες καταργώντας ε, την ασυλία εκατοντάδων βουλευτών δεν μπορεί να γίνεται λόγος λοιπόν για την ε, θεσμική σταθεροποίηση. Για την προστασία μειονοτήτων ούτε και για αυτή μπορεί να γίνεται λόγος διότι εδώ στρέφονται αυτά τα μέτρα κατά της κουρδικής μειονότητας. Για την κοινοβουλευτική δημοκρατία όποιος εκλέγεται πρέπει να έχει την δυνατότητα και το δικαίωμα να ασκεί το αξίωμά του αυτό χωρίς να διώκεται, χωρίς να απειλείται με διώξεις. Ας δούμε τα άλλα θεσμικά όργανα στην Τουρκία. Τι γίνεται με αυτά τότε βλέπουμε ότι σε σχέση με την εισαγγελία ότι το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο έχει διαπιστώσει ότι πρόκειται για πολιτική δικαιοσύνη και όχι για ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Αν δούμε τι γίνεται με τα μέσα του τύπου, με την δίωξη εφημερίδων και δημοσιογράφων από το καθεστώς Ερντογάν, όταν βλέπουμε ότι απειλείται η ελευθερία του συναθρίζεστε, αλλά και κοινωνικών ομάδων που διώκονται όταν το, ε, ο στρατός ε, δεν περιορίζεται αλλά ίσα ίσα επιβάλλει τις, ε, τις διώξεις σε άλλους. Όταν βλέπουμε ότι διώκεται το ΧΑΝΤΕΠΕ τότε πρέπει να τεθεί το ερώτημα η κατάσταση ασφάλειας στην Τουρκία βελτιώνεται ή όχι. Το αντίθετο συμβαίνει, επιδεινώνεται και αυτό είναι αντιπαραγωγικό και όχι μόνο υπό το πρίσμα της Ευρώπης αλλά και υπό το πρίσμα των πολιτών της Τουρκίας. Σήμερα, παρακαλώ στη συνέχεια. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, ένας χρόνος πέρασε από τότε που η ΧΑΝΤΕΠΕ σημείωσε μια εκλογική νίκη 7 Ιουνίου πέρυσι. Στις 7 Ιουνίου ακριβώς ο Ερντογάν υπέγραψε το νόμο που θα οδηγήσει στην άρση ασυλίας εκατοντάδων βουλευτών της Μεγάλης Τουρκικής Εθνοσυνέλευσης. Και αυτό ακριβώς το γεγονός δεν είναι πλέον κάτι το τυπικό ως παράπτωμα του Προέδρου, αλλά ένα συνειδητό βήμα του Προέδρου προς ένα προεδρικό αυταρχικό σύστημα το οποίο θα επιβληθεί η εκπροσώπηση με την επιβολή των ε, κελευσμάτων του κόμματος ΑΚΠ βλάπτει την τουρκική δημοκρατία. Αυτός ο νόμος έχει όμως και επιπτώσεις στους ίδιους τους βουλευτές στην άσκηση του έργου τους, ε, του αξιώματός τους. Ε, μένουμε πραγματικά με το στόμα ανοιχτό στην Ευρώπη πώς με τέτοιο τρόπο δημιουργείται ένα κλίμα φόβου και ένα κλίμα διώξεων στην Τουρκία και αυτό δεν στρέφεται μόνο κατά των βουλευτών της ΧΑΝΤΕΠΕ. Αν δούμε το παράλογο της υπόθεσης ότι λόγω του ότι υιοθετήθηκε ένα ψήφισμα στην Ομοσπονδιακή Βουλή της Γερμανίας. Τώρα ζητεί ο Ερντογάν να γίνονται αιματολογικοί έλεγχοι βουλευτών του ε, Γερμανικού Κοινοβουλίου τουρκικής ε, καταγωγής. Όλα αυτά, επειδή αυτοί ενέκριναν ένα τέτοιο ψήφισμα, όλα αυτά δείχνουν ότι δίνει μάχη ο Ερντογάν στα, κατά των δικαιωμάτων ελεύθερης έκφρασης των βουλευτών. Και αυτό, αν γινόταν εδώ, τότε τρία τέταρτα των Ευρωβουλευτών πραγματικά θα ε, στερούντο την ασυλία τους και τα δικαιώματά τους, διότι πρόκειται πραγματικά για ένα πλήγμα κατά της ελευθερίας και της ελευθερίας της έκφρασης. Και θέλω να πω ότι σε σχέση με τους 59 βουλευτές της ΧΑΝΤΕΠΕ βρίσκονται και δύο που γνωρίζουμε πολύ καλά στο Ευρωκοινοβούλιο. Η Λέιλα Ζανά αφενός που πήρε το βραβείο Σαχάροφ ε, από το Ευρωκοινοβούλιο και που ακριβώς έδωσε μάχη για την ελευθερία της έκφρασης και πήρε αυτό το βραβείο. Και η Φέλεκνες Ούτσα που πάλι ε, είναι γνωστή για το ότι έμαθε τα ε, όσα αφορούν τη δημοκρατία εδώ και τα μετέφερε στην Τουρκία και δεν μπορούμε να δεχθούμε την ε, δίωξη αυτών των προσωπικότητων και πρόκειται και για πολύ περισσότερους και περισσότερα ακόμα και όταν λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι, πρέπει, ότι έχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη λέει, ε, πρέπει να πούμε ότι 228 ε, δικαστές και εισαγγελείς μετατέθηκαν από το καθεστώς ε, Ερντογάν. Πώς είναι δυνατόν να υπάρχει λοιπόν εμπιστοσύνη σε ένα τέτοιο καθεστώς και σε μια τέτοια δικαιοσύνη. Ένας άλλος τρόπος προσέγγισης χρειάζεται εδώ και πρέπει πραγματικά να δράσουμε ώστε από κοινού να προστατεύσουμε την ευρωπαϊκή ελευθερία και δικαιοσύνη δικαιοσύνη. Ευχαριστώ. Βαλέρο παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είναι επικίνδυνο να εκλεγεί κανεί ε, στην τουρκική εθνοσυνέλευση γιατί μπορεί να μπει φυλακή. Παρά το ότι είναι δύσκολο να εκλεγεί γιατί υπάρχει 10% κατόφλιο. Παρόλα αυτά, ε, ορισμένοι κατάφεραν να δημιουργήσουν ένα συνασπισμό για να μπορέσουν να ε, εκλεγούν. Και παρά το ότι στις τελευταίες εκλογές ε, πήραν μικρότερο ποσοστό, παρόλα αυτά μπήκαν και πάλι στη Βουλή. Η έκθεση πρόοδου της Κομισιόν για τις τελευταίες εκλογές λέει ότι υπάρχει ε, παρενόχληση και πιέσει και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα κόμματα τη αντιπολίτευσης και μία ατμόσφαιρα απειλών και βία κατά των υποψηφίων και επιδρομές στα γραφεία των κομμάτων τη αντιπολίτευσης και ε, το ΧΑΝΤΕΠΕ το έχει υποστεί αυτό και άλλα κόμματα και πρόσφατα το Κοινοβούλιο το περασμένο, μα αυτό το μήνα ενέκρινε ένα νόμο που επιτρέπει διώξει κατά των βουλευτών που θεωρούνται ε, μπορούν να θεωρηθούν λοιπόν υπεύθυνοι για εγκλήματα κατά του τουρκικού κράτους. Ε, ενώ εμείς συζητάμε απελευθέρωση των θεωρήσεων. Πρέπει να σκεφτούμε ε, εάν λαμβάνουμε υπόψη αρκετά την ελευθερία του τύπου, την ελευθερία της έκφρασης και πόσοι από εμά ανοιχτά επικρίνουμε τον Τούρκο πρόεδρο. Πόσοι από εμά θα ήμασταν φυλακοί αν ήμασταν Τούρκοι πολίτες. Πόσοι από εμά δεν θα ε, είχαμε υπογράψει δηλώσεις όπως αυτές των πανεπιστημιακών κτλ. Ε, ξέρουμε ότι έχει αρθεί η ασυλία. Μήπως θα έπρεπε να αρθεί και για τον ίδιο τον πρόεδρο με αυτά που γίνονται ή για αυτούς που ψηφίζουν τέτοια πράγματα. Είναι απαράδεκτο αυτό και δεν μπορεί να θεωρήσει η Τουρκία ότι με αυτόν τον τρόπο θα υπάρξει φιλελευθερωποίηση των ε, θεωρήσεων. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα εκφράσει τις ανησυχίες, του, τις ανησυχίες του για τον πολύ ασαφή ορισμό της τρομοκρατίας, του οργανωσμένου εγκλήματος και της προπαγάνδας κατά του κράτους. Είναι πολύ δύσκολο να καθοριστούν επακριβώς τα αδικήματα που περιλαμβάνονται σε τόσο ευρύς ορισμούς. Και επίσης διαπιστώνουμε ότι μετά τα προβλήματα διαφθοράς του 2013 ε, ο Πρόεδρος ε, έχει αποκτήσει όλο και περισσότερη εξουσία και κάνει όλο και πιο δραστικούς ε, αντιτρομοκρατικούς νόμους οι δικαστές, οι μειονότητες, οι πανεπιστημιακοί, οι δημοσιογράφοι όλοι αυτοί υφίστανται διώξεις. Ο Ερντοάν θα έπρεπε να τρέπεται για αυτά τα οποία εγκρίνει. Ο κ. για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πραγματικά για ποιο λόγο να ψηφίζει κανείς αυτή τη στιγμή στην Τουρκία, τη στιγμή που βλέπουμε να προκύπτουν όλες αυτές οι εξελίξεις. Μια εξέλιξη η οποία στρέφεται κατά των ίδιων των βουλευτών και ιδίω των βουλευτών του ΧΑΝΤΕΠΕ. Βλέπετε αυτή τη στιγμή ότι τα δεδομένα θα αλλάξουν στο τουρκικό κοινοβούλιο. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, ο Ερντογάν θέλει να αλλάξει εντελώ το σύνταγμα τη χώρα προκειμένου να ανακτήσει περισσότερε εξουσίε. 138 Κούρδοι βουλευτές αυτή τη στιγμή κινδυνεύουν από τη νέα αυτή απόφαση και βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι η κατάσταση είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολη. Αν δείτε τα νέα τα οποία μας φτάνουν καθημερινά από την Άγκυρα. Πρόκειται για μία ακόμα πράξη στην οποία προχωρά ο Ερντογάν απέναντι σε μια Ευρώπη η οποία δεν έχει το θάρρο να καταγγείλει τι πράξει αυτέ του Ερντογάν. Πώ μπορούμε εμεί να μιλάμε αυτή τη στιγμή για διαδικασία προσχώρηση με αυτή τη συγκεκριμένη Τουρκία που καταπατά τα δικαιώματα των βουλευτών δεν μπορούμε να αποδεχθούμε την πράξη αυτή, την άρση των βουλευτών. Το πρόβλημα δεν είναι το ότι καταστέλει ο Ερντογάν τη δημοκρατία, αλλά ότι εμεί σιωπούμε ω Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα λεπτό, κύριο Σφερό. Όλο περισσότερα κάνετε, κύριε Ερντογάν. Μέχρι πότε, μετά τον εκβιασμό για του μετανάστε, να άλλη μια προσπάθεια ε, από τον Ερντοάν που θέλει να καταργήσει την ε, αντιπολίτευση. Έναν αιώνα μετά την γενοκτονία κατά των ε, Κούρδων και των ε, Ασυρίων καμία προσπάθεια από πλευρά της Ευρώπης. Τι διαπιστώνουμε, ότι η Τουρκία απειλεί την Ευρώπη. Η ομάδα μας, η Ευρώπη των Εθνών, σας έχει θέσει ενώπιον των ευθυνών σας. Τι περιμένετε αγαπητοί συνάδελφοι, τι, τι περιμένετε για να ζητήσετε τη διακοπή των διαπραγματεύσεων ένταξη. Θεωρείτε ότι η δικτατορία του Ερντοάν είναι πρότυπο ε, που συνάδει με τις αξίες μα. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Συναδεινός, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, πρόσφατα ο Κούρδος βουλευτής της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, Ενκούφερ Χατ, δήλωσε με θάρρος ότι η Τουρκία δεν είναι τίποτα παρακλεμένη γη Ελλήνων, Αρμενίων και Κούρδων. Όπως είπε, μάρτης μου η ιστορία. Συνεχίζοντας την παράθεση παραδειγμάτων για τις αποτρόπες πράξεις των Τούρκων, είπε «Εμείς οι Κούρδοι ζούμε στο Κουρδιστάν και όταν ζούσαμε σε αυτή τη γη οι τούρκοι ήσαν στη μογγολία απασχολημένοι με τα άλογά τους αυτή δε η γη μας ανήκει και μένουμε εδώ. η σύγχρονη τουρκία είναι μικρότερη των 100 ετών ενώ το κουρδιστάν είναι άνω των 5.000 ετών και υπάρχουν δεκάδες αρχαία ελληνικά κείμενα που αναφέρουν το όνομα των Κούρδων και του Κουρδιστάν. Σας διαβάζω μερικές από τις απειλές των Τούρκων βουλευτών μελών του Κοινοβουλίου. Φυτέψτε του μια σφαίρα στο κεφάλι. Πυροβολήστε τον. Υπέγραψε τη θανατική σου καταδίκη. Το κεφάλι σου θα κυλήσει αλήτη Κούρδε. Βάλτε τον φυλακή για δέκα χρόνια. Θα καταστρέψουμε τι πόλεις σα. Θα ήθελα να ρωτήσω βέβαια τον κύριο Σούλτς σε ποιον θα επέβαλε τι κυρώσει που πρόσφατα επέβαλε σε μένα. Στο θαραλέο Κούρδο βουλευτή ή στους αντίστοιχους Τούρκους. Στην κοινοβουλευτική δημοκρατία που θεσμικά ο πρόεδρος προστατεύει, τι είναι άραγε πιο κατακριτέα. Η στάση τουρκου στην Κούρδου που θεσμικα ο προεδρο προστατευει τι ειναι αραγε πιο κατακριτεα η σταση του κουρδου που επικαλεστηκε την ιστορική αλήθεια ή των Τούρκων που τον έβρισαν του απείλησαν τη ζωή και διαπράττουν εγκλήματα κατά αμάχων. τελευταία δε δεν σεβάστηκαν ούτε το θρησκευτικό μνημείο της αγίας σοφίας. τα παραπάνω τα αφιερώνω στον αγαπητό πρόεδρο για τους προστατευόμενους του τούρκους που σαν πρώην βιβλιοπόλης έπρεπε να γνωρίζει καλώ την ιστορία για να λαμβάνει δίκαιες αποφάσεις. ευχαριστώ. Ε, Ένα λεπτό κυρία Ζώμα καταπατά όλα τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η άρση τη ασυλίας ενό τετάρτου των βουλευτών τη μεγάλη τουρκική Εθνοσυνέλευση είναι άλλο ένα ράπισμα κατά τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ και πολύ καιρό οι επικριτέ του καθεστώτο αντιμετωπίζονται ως τρομοκράτες και καταδικάζονται σε ε, μακροχρόνιε ε, ποινέ φυλάκιση. Και τώρα αυτό φαίνεται ότι θα αντιμετωπίζει και η τουρκική αντιπολίτευση στο Κοινοβούλιο που πρέπει να εξαλειφθεί από ό,τι φαίνεται. Και θα εξαλειφθεί. Έτσι θα απελευθερωθεί ο δρόμος για νέες εκλογές όπου οπωσδήποτε το ΑΚΠ θα πάρει ε, τις αναγκαίες έδρες για να μπορέσει να κάνει συνταγματική μεταρρύθμιση και να κάνει προεδρική δικτατορία τη χώρα ο Ερντοάν Είναι δράμα αυτό για τη χώρα που υπάρχει εδώ και πολύ καιρό κλίμα φόβου. Αλλά είναι μεγάλο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί χρειαζόμαστε ε, αξιόπιστου εταίρου. Γιατί πρέπει να συνεργαστούμε με την Τουρκία. Αλλά η χώρα δεν είναι πλέον αξιόπιστη, δεν είναι υπεύθυνη. Πρέπει λοιπόν να αντιδράσουμε. Πρέπει επιτέλους και τελειωτικά να διακόψουμε τις ενταξιακές διαπραγματεύσεις. Ο κύριος ένα λεπτό. Αρχικά θα ήθελα να εκφράσω τα συλληπιτήριά μου για τα θύματα των πρόσφατων τρομοκρατικών επιθέσεων στην Τουρκία. Φίλε και φίλοι, ο κύριος Ερντογάν οδηγεί την Τουρκία σε πολιτικό μεσαίωνα το αποτέλεσμα των επιλογών του των πολιτικών του επιλογών τον πληρώνει καθημερινά ο τουρκικό λαό. Άρει την ασυλία των βουλευτών του ΧΑΝΤΕΠΕ με την κατηγορία ότι στηρίζουν την τρομοκρατία. Δεν μπορούμε να παραμένουμε απλοί θεατέ στη δίωξη βουλευτών μόνο και μόνο επειδή είναι Κούρδοι. Δεν γίνεται να μένουμε απαθεί σε σφαγέ πολιτών και καταστροφέ ολόκληρων πόλεων όπω είναι ο Σαϊμπίν. Συγχρόνω απειλεί Γερμανού βουλευτέ τουρκική καταγωγή που ψήφισαν την αναγνώριση τη γενοκτονία των Αρμενίων τέλος προσβάλλει την αγία σοφία ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς σύμβολο του χριστιανισμού χρησιμοποιώντας το για φθηνή προπαγάνδα. όλα αυτά είναι εχθρικά προς ευρωπαϊκές αξίες της δημοκρατίας του πολιτισμού και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. οφείλουμε λοιπόν όλοι μαζί σήμερα να στείλουμε ένα ηχηρό μήνυμα ότι ο κύριος ερντογάν είναι αυτός που κλείνει την πόρτα της ευρωπαϊκής προοπτικής για τη χώρα του την τουρκία. Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριο Ντεμεσμάκερ έχει το λόγο για 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Σα άκουσα με ιδιαίτερα ενδιαφέρον και συνειδητοποιώ ότι ενισχύετε πάρα πολύ για την κατάσταση και ότι θα επιληφθείτε όντω τη κατάσταση αυτή. Εγώ ανησυχώ πάρα πολύ για το πόσο ρεαλιστική τελικά είναι στη στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί από ό,τι φαίνεται δεν συντοπεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή μονοπολεί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και προσπαθεί μέσω των πράξεων αυτών να βάλει κατά του ίδιου του Κουρδιστάν και βέβαια των βουλευτών από την περιοχή αυτή. 138 βουλευτές κινδυνεύουν με άρση της βουλευτικής ασυλίας. Καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε για ανθρώπους που έχουν εκλεγεί δημοκρατικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, θεωρώ. Ή είμαστε αρκετά διπρόσωποι απέναντι στην Τουρκία. Και αυτό είναι πολύ λανθασμένη στάση. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, θα ήθελα να γνωρίζω πολύ καλά ποια είναι η στάση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μα λέτε ότι ανησυχείτε πολύ και ότι πρέπει να παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά την κατάσταση. Ε, αυτό δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Πόσο θα συνεχίζουμε να είμαστε όμοιροι της Τουρκίας. Πότε θα συνεχιζουμε να ειμαστε ομοιροι τη τουρκια ποτε θα σταθουμε απεναντι στον Ερντογάν λέγοντά του ότι η Συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση και Τουρκία για το μεταναστευτικό δεν είναι λευκή επιταγή και ότι σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε εμεί στο όνομα τη συμφωνία αυτή να αποδεχθούμε την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η κυρία Σάκη, για ένα λεπτό παρακαλώ. Το μικρόφωνο σας παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Είδαμε απαράδεκτες συμβιβασμούς από πλευράς κομισιών και κρατών μελών για τις αξίες πάνω στις οποίες έχει οικοδομηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ελπίζουν ότι η Τουρκία θα, προσπαθήσει, θα προστατεύσει τα σύνορά μας. Το θέμα είναι πότε θα φέρει αποτελέσματα. Η Ευρώπη έχει συμφωνήσει το 2013 72 κριτήρια με την Ευρώπη. Το θέμα είναι ότι πρέπει η τρομοκρατία να αντιμετωπιστεί αλλά θα πρέπει να μπορούν οι Τούρκοι βουλευτές να εκπροσωπήσουν δημοκρατικά τους ε, ψηφοφόρους τους. Η μαζική άρση ασυλίας δεν είναι δέουσα σωστή ε, διαδικασία. Μιλήσατε κύριε Επίτροπε για τη σημασία του κράτους δικαίου. Σας κάνω έκκληση να εξασφαλίσουμε ότι εμείς η Ευρωπαϊκή Ένωση θα κινηθούμε με βάση το διεθνές δίκαιο και θα εξασφαλίσουμε ότι η Τουρκία θα κάνει το ίδιο. Δεν θέλουμε περαιτέρω συμβιβασμούς ούτε στο πλαίσιο της συμφωνίας για το μεταναστευτικό ούτε για την ενίσχυση της αντιτομοκρατικής νομοθεσίας και βεβαίως θέλουμε να είμαστε ηγέτες στον κόσμο. Επόμενος ομιλητής ο κύριος Χατζηγεωργίου για ένα λεπτό. Θέλω και εγώ να εκφράσω τα συλληπιτήριά μας για τους νεκρούς της χθεσινής βομβιστικής επίθεσης γιατί καμιά εξήγηση δεν μπορεί να δοθεί σε τέτοιες βάρβαρες πράξεις. Όμως και οι ενέργειες του κυρίου Ερτογάν είναι βόμβα μεγατόνων στα θεμέλια της τουρκικής δημοκρατίας. Ήδη μετράμε 300.000 εκτοπισμένους Κούρδους από τα σπίτια τους και στόχο των ενεργειών του όσον αφορά την άρση τη ασυλία των Κούρδων βουλευτών είναι η υποταγή του κούρδικου πληθυσμού. Μπροστά σε αυτό νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δείξει την αξιοπρέπειά τη πρώτα απ' όλα απέναντι στον εαυτό τη. Πρώτα απ' όλα απέναντι σε εμά δεν πρέπει να επιτρέψουμε να δώσουμε την εντύπωση ότι υποτασσόμαστε μπροστά στο γεγονό ότι η Τουρκία φιλοξενεί τα τρία εκατομμύρια των προσφύγων και αξιοποιεί ή εκμεταλλεύεται τόσο πολύ καθαρά αυτό το γεγονό απέναντι στο σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών. πρέπει να δοθεί καθαρό μήνυμα στον τούρκο πρόεδρο ότι θεωρούμε τις πράξεις του ότι ανατινάσουν τις σχέσεις του με την ευρωπαϊκή ένωση. ευχαριστώ. Η κυρία Κέλλερ, Κέλλερ ευχαριστώ. Η άρση της ασυλίας είναι, ε, στοχεύει κατά των ε, βουλευτών του ΧΑΝΤΕΠΕ και είναι σαφής και η πρόθεση θέλει να κάνει το HDP να σιωπήσει και το κόμμα HDP να σιωπήσει. Αυτό είναι εντελώ αντιδημοκρατικό. Ποινικοποιεί ένα ολόκληρο κόμμα που εκπροσωπεί ένα ε, σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, του εκλογικού σώματος. Και δεν ψήφισαν μόνο οι Κούρδοι για το ΧΑΝΤΕΠΕ. Πολλοί που πίστευαν σε ένα διαφορετικό μέλλον για την Τουρκία το ψήφισαν πολλοί που ήθελαν να διαμαρτυρηθούν για τις επιθέσεις κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κατά τη ελευθερία του τύπου, όλα αυτά τα οποία εκπροσωπούμε. Πρέπει λοιπόν να τους στηρίξουμε. Είναι έσχος το ότι έχει ξεσπάσει και πάλι ο, ο πόλεμος στο Κουρδιστάν. Και είναι κρίμα, διότι ο Ερντοάν ε, είχε κάνει αρκετά βήματα προ την προσπάθεια μια βιώσιμη λύση. Αλλά τώρα έχουμε επανέλθει στο, στην αφετηρία, Χιλιάδες ε, άμαχοι έχουν ε, ε, θανατωθεί, έχουν πεθάνει και ολόκληρες πόλεις ισοπεδώνονται. Άρα έχουμε μια τρομερή απώλεια, την απώλεια της ίδιας της ειρηνευτικής προσπάθειας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε πολύ στεναρή αντίδραση. Πρέπει να εκφράσουμε σαφώς τις αξίες μας. Δεν μπορούμε να σιωπούμε όταν αυτοί που προσπαθούν να εκφραστούν αναγκάζονται σε σιωπή, φημώνονται. Έχουμε κάνει πολλά λάθη στο παρελθόν ως Ένωση, αλλά και τα κράτη-μέλη. Στην ουσία ε, ενισχύσαμε τον Ερντοάν. Δεν πρέπει να επαναλάβουμε αυτά τα λάθη. Πρέπει να στρίξουμε αυτούς που υπερασπίζονται τις αξίες μας. Μόνο έτσι θα βοηθήσουμε να υπάρξει μια καλύτερη Τουρκία. Η κυρία Όμπερμαϊρ, ένα λεπτό. Ο κύριος Όμπερμαϊρ. Ευχαριστώ. Από ό,τι λέγεται, ε, από ό,τι είπε ο Ερντοάν, στις 20 Μαΐου θα πρέπει να πληρώσουν οποιαδήποτε τιμή αυτοί οι βουλευτές. Αλλά αντί να αντιδράσετε όπως πρέπει κύριε Χάν, ε, συνάπτουμε συμφωνίες με αυτόν τον άνθρωπο και αγνοούμε το γεγονός ότι διαλύει τη δημοκρατία αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Τους υποσχόμεθα δισεκατομμύρια, κεφάλαια, ότι θα ανοίξουμε, διευκόλυνση για τις θεωρήσεις. Ε, μας κοροϊδεύει ο Ερντοάν και μόνο, μόνο και μόνο για να, για να σώσουμε το κεφάλι το πολιτικό μέλλον δηλαδή της Μέρκελ και οδηγούμε ολόκληρη την Ευρώπη στην καταστροφή. Και επιπλέον ο Έρντοαν μας ε, απειλεί με εκατομμύρια νέων προσφύγων και ότι θα κινητοποιήσει τους Τούρκους που ζουν στη Γερμανία εναντίον μας. Και δεν είναι δυνατόν να δεχόμαστε να αντιδρούν έτσι όταν δεν θέλουμε να σιωπήσουμε και για την γενοκτονία των ε, Αρμενίων. Πρέπει να ξυπνήσει η Ευρώπη. Κόρβιν Μίκε, 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Ένας βουλευτής, μία, ε, μία ε, τουρκάλα βουλευτής καταδικάστηκε σε ισόβια αλλά τελικά την πήγανε ε, με ειδικά μέσα στο, στη Μεγάλη Βρετανία επειδή ήταν βουλευτής εδώ και μερικέ δεκαετίε ο Χίτλερ ήταν αυτό ο οποίο αφαίρεσε τα δικαιώματα από του βουλευτέ τη αντιπολίτευση, ε, μερικού μόνο μήνε μετά ε, από την ε, ανάληψη εξουσία για την οποία τα κόμματα τη αντιπολίτευση δεν είχαν αντιδράσει όπω έπρεπε. Ο κύριο Ερντοάν έχει ήδη καταστρέψει δύο κόμματα τη αντιπολίτευση. έχει τώρα την πλειοψηφία που θα το επιτρέψει να κάνει ό,τι ακριβώ γουστάρει. Και τα δύο κόμματα που υποστήριξαν, που τον υποστήριξαν σε αυτή την επιλογή και αυτά τελικά θα το μετανιώσουν. Τώρα το θέμα που τίθεται είναι γιατί εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζουμε τον κύριο Ερντοάν. Ε, παρακαλώ δώστε μου μια απάντηση. Ήδη έχει πάρει τρία δις. Φαίνεται ότι ορισμένα από αυτά τα τρία δί τα έδωσε πίσω σε ορισμένους από τους Ευρωπαίους που διαπραγματεύονται μαζί του. Μόνο αυτή την απάντηση μπορώ να δώσω εγώ σε αυτά που συμβαίνουν. Τελικά η δεξιοτεχνία της κυρίας Μέρκελ είναι μικρότερη από ό,τι ε, θεωρούμε και οι Γερμανοί βουλευτέ έλαβαν τη σωστή απόφαση παρά τι πιέσει τη. Μα έδειξαν τον δρόμο. Όσοι υποκλίνονται μπροστά στον Ερντοάν είναι απειλή για όλη την Ευρώπη. Γιατί η Τουρκία θα συνεχίσει να απειλεί την Ευρώπη ολόκληρη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Σόντροβα έχει το λόγο για ένα λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Νομίζω ότι ε, σήμερα η ανταπόκρισή σας ήταν ανεπαρκής. Αυτό που θα περίμενα εγώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να απορρίψει ρητός και σαφώς όλες αυτές τις πράξεις ε, του ε, τουρκού προέδρου που ουσιαστικά φημώνουν ε, την ελευθερία της έκφρασης και γενικότερα καταπατούν τη δημοκρατία στην Τουρκία. Και υπάρχει και η περίφημη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας. Ας μην το ξεχνάμε αυτό. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι φαίνεται, είναι ξεκάθαρο ότι ο Ερντογάν στρέφεται κατά συγκεκριμένων βουλευτών από το ΧΑΝΤΕΠΕ, και είναι επονίδιστη και στάση του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ε, του ΤΣΕΧΑΠΕ. Αν πραγματικά η Τουρκία θέλει να έχει ελευθερία όσον αφορά μάλλον την απελευθέρωση των θεωρήσεων, τότε θα πρέπει πραγματικά να σέβεται το κράτος δικαίου και τα δικαιώματα των πολιτών και των βουλευτών. Διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να συνεχίσει να πραγματεύεται για απελευθέρωση των θεωρήσεων. Ευχαριστούμε. Έχετε από τον κύριο Σόνιν μια μπλε κάρτα. Τη δέχεστε. Παρακαλώ. Κύριε Σόνιγκ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Απευθύνομαι σε εσά, κυρία Σόιντροβα. Πήρατε το λόγο και στέλνετε αυτή τη στιγμή ένα πολύ ηχηρό μήνυμα με το οποίο συμφωνώ. Όντω, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι πήραν το λόγο και στείλανε ένα πολύ ηχηρό μήνυμα απέναντι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και την Τουρκία. Υπάρχει όμω ένα κράτο τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ουγγαρία, με επικεφαλή τον κύριο Ορμπάν, ο οποίο αναφέρθηκε ως υποδειγματικός ηγέτης και από τον Πούτιν και από τον Ερντογάν. Η δική σας η πολιτική ομάδα πότε επιτέλους θα ανταποκριθεί στις δηλώσεις αυτές, γιατί στη δική σας πολιτική ομάδα νίκη ο κύριος Όρμπαν. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να απαντήσω στην ερώτηση του συναδέλφου Κατά την άποψή μου, ο κύριος Πούτιν δεν αποτελεί παράδειγμα που θα πρέπει να ακολουθούμε και ο κύριος Ερντογάν από την άλλη δεν αποτελεί ούτε και αυτός υπόδειγμα, γιατί περιορίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα πολιτικά δικαιώματα και τη δημοκρατία. Ευχαριστούμε πολύ ο κύριος Βάλτεν Χόρζερ. Αγαπητοί συνάδελφοι, η κοινοβουλευτική ασυλία είναι πολύτιμο αγαθό που πρέπει να υπάρξει σε οποιαδήποτε δημοκρατία. Η άρση της πρέπει να γίνεται μόνο σε κατεξαίρεση καταστάσει και μπορεί να γίνει μόνο μεμονωμένα μετά από εξέταση των περιστάσεων. Τα γεγονότα των τελευταίων ημερών είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά γιατί είναι συλλογική κύρωση και μεταξύ των τιμωρωμένων υπάρχουν γνωστοί. Ο κύριο Ντεμιρτά, που πριν από μερικέ εβδομάδε ήταν προσκεκλημένος στους σοσιαλιστέ και ο Φελίκνα Ούκα που ήταν 10 ε, χρόνια ευρωβουλευτή. Είναι παράλογο αυτά που γίνονται. Αυτοί οι συνάδελφοι φυσικά δεν είναι αντικείμενο, δεν μπορεί να είναι αντικείμενο υποψιών. Έχουμε συζητήσει συχνά μαζί του και ξέρουμε ότι πάντα εκφράζονταν υπέρ μια ειρηνική λύσης του κουρδικού θέματος. Ο κύριος Τσάρλ Τάνοκ, 1,5 λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, η άρση της ασυλίας από πολιτικούς και η ποινικοποίηση τη δραστηριότητά του θα το καλωσορίζαμε σε μια δημοκρατία. Όμως οι διαδικασίες ε, φαίνεται ότι έχουν πολιτικούς λόγους. Είναι μια συλλογική κύρωση για να αποδυναμώσει την, ε, το κόμμα Χαντεπέ που έχει κουρδική πλειοψηφία διότι ο Έρντοκαν θεωρεί ότι είναι υποκατάστατο του, του ΠΚΚ με το οποίο έχει πόλεμο στην Ανατολική Τουρκία και θέλει να έχει ανεξέλεγκτες προεδρικές εξουσίες για να έχει το αναγκαίο επίπεδο εξουσιών του ε, πρόσφατα οικοδομημένου ε, παλατιού του που είναι σαν ε, παλάτι Σουλτάνου και για να έχει την αναγκαία κοινοβουλευτική πλειοψηφία για συνταγματική μεταρρύθμιση κάνει ό,τι μπορεί. Και τον άτακτο πρωθυπουργό του τον έδιωξε και προσπαθεί τώρα να βρει υποστήριξη και εκτός του κόμματο του. επειδή μειώνεται μετά από 20 χρόνια η εξουσία του επικεφαλής του ΜΕΧΑΠΕ φαίνεται ότι έκανε μία συμφωνία με τον πρώην ε, αντίπαλό του Μπαχτσέλη για να λάβει την ε, δική του στήριξη στην μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση. Άρα απειλείται και η δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Και αυτές είναι απλώς οι τελευταίες εξελίξεις σε μια ευρύτερη προσπάθεια, ένα ευρύτερο εγχείρημα για να ε, ε επιβληθούν οι στόχοι του ΑΚΠ. Φυσικά έχει μεγάλη αξία η Τουρκία για την Ένωση ως υποψήφια χώρα και είναι σύμμαχός μας στο ΝΑΤΟ και είναι αναγκαίος ο μας για να σταματήσει ο ροή προσφύγων από τη Συρία. Αλλά ο Ερντοάν μετατρέπει τη χώρα του που δεν είναι η δημοκρατία πριν από 20 χρόνια και όλοι θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα ανήσυχοι γι' αυτό. Βάγγελ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Η απόφαση αυτή για την άρση της βουλευτικής ασυλίας κατά των βουλευτών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης κατηγορώντας τους για διάφορα πράγματα, εικασίες, για συνωμοσίε κτλ. Τα έχουμε δει και στο παρελθόν. Ουσιαστικά ο Ερντογάν θέλει να συγκεντρώσει στο πρόσωπό του όλη την εξουσία. Αυτό βλέπουμε τα τελευταία χρόνια και αυτό βλέπουμε αυτή τη στιγμή με το στρατηγικό μας εταίρο την Τουρκία. Και το αποκορύφωμα ήταν βέβαια η απόφαση αυτή για την άρση τη βουλευτική ασυλία, την οποία την καταγγέλουμε προφανώ. Χρειαζόμαστε την Τουρκία. Η Τουρκία πλήττεται από την τρομοκρατία και αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στην όλη περιφέρεια. Και βέβαια το χειρότερο ενδεχόμενο είναι ακριβώς αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Το να οδηγηθεί ο Ερντογάν σε αποφάσεις οι οποίες είναι απολυταρχικές. Πραγματικά μπορούμε να δεχθούμε ένα τέτοιο καθεστώς στην Τουρκία. Μπορούμε να καταλήξουμε σε κοινά συμφέροντα και κοινέ αξίες. Κυρία Merci, Monsieur le Président. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χτες, ακριβώς ένα χρόνο μετά τις ε, από τις κοινοβουλευτικές εκλογές, ο Ρατζή Περτογάν ήρε συλλογικά την ασυλία 135 βουλευτών, εκ των οποίων 103 από το ε, κόμμα, το φιλοκουρδικό κόμμα αρέσουν στον κύριο Ερντογάν τα σύμβολα, αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε πλέον αυτό το αυταρχικό καθεστώς. Πολλά έχουν αλλάξει. Πρέπει μια χώρα υποψήφιο να ε, τηρεί τις δημοκρατικές αρχές, αλλά αυτό φαίνεται να μην απασχολεί τον ε, πρόεδρο της Τουρκίας με την πράξη του εναντίον του Αστομπέκ μπορεί οι βουλευτές να ξαναβρεθούν στη φυλακή. Εδώ διακυβεύεται η ελευθερία της έκφρασης. Ως βουλευτές δεν μπορούμε να παραμείνουμε σιωπηλοί. Κάνω επίσημα έκκληση στην αλληλεγγύη ώστε ε, ο καθένας μας να στηρίξει ατομικά τους βουλευτές. Πρέπει να δείξουμε μια ισχυρή πολιτική. Ο κύριος Μαραγάλη ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Χθε ε, έκλεισε χρόνος από τις εκλογές και για πρώτη φορά τότε πριν από ένα χρόνο ο κουρδικό κόμμα είχε μπει στη Βουλή με 13% των ψήφων. Και ένα χρόνο μετά μετά από μια καμπάνια συκοφάντησης του κόμματο και μετά τις νέες εκλογές του Νοεμβρίου η κατάσταση έχει αλλάξει 180 μοίρε. Ο πρόεδρο Ερντοάλ υπέγραψε τον νόμο τη συνταγματική μεταρρύθμιση που του επιτρέπει να άρει την ε, νομοθετική ασυλία. Πρώτη επίπτωση, τουλάχιστον 50 βουλευτέ ε, Κούρδοι κινδυνεύουν ε, με καταδίκες και φυλακίσεις για την απλή έκφραση των πεπιθήσεών τους. Έχει περάσει ένας χρόνος Τότε, πριν από ένα χρόνο, η κατάσταση ήταν πολύ θετική και υπήρχε εμπλοκή της ε, κοινωνίας. Αλλά τώρα η κατάσταση είναι τρομερή, υπάρχει σοβαρή αντιδημοκρατική εξέλιξη και τρομερή σύγκρουση. Είναι σαφές οι δύο λύσεις. Ή ε, αυταρχισμός ή δημοκρατία. Μόνο η τελευταία λύση εξυπηρετεί τα συμφέροντα της τουρκικής κοινωνίας. Πρέπει να προωθήσουμε μία ε, δημοκρατική εναλλακτική λύση. Ο κύριος Επιτίδος ένα λεπτό λέει ο πρόεδρος. Ένα λεπτό και 30 δευτερόλεπτα. Ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ε, πριν ε, μερικές μόλις ημέρες το τουρκικό κοινοβούλιο ενέκρινε την άρση της ασυλίας 138 βουλευτών μεταξύ των οποίων 103 του ΧΑΝΤΕΠΕ του φιλοκουρδικού κόμματος το οποίο είναι και η τρίτη πολιτική δύναμη της χώρας το έγκλημα το οποίο έκαναν οι βουλευτέ αυτοί ήταν ότι ζητούσαν να σταματήσουν οι επιχειρήσει των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων στην νοτιοανατολική τουρκία εναντίον των κούρδων και να αρχίσουν οι ειρηνευτικές συνομιλίε και πάλι. παρ' όλα αυτά ο πρόεδρος ερντογάν τους ε, κατήγγειλε και τους εδίωξε με βάση τον νόμο κατά τη τρομοκρατία. με σκοπό να του κλείσει στη φυλακή και να μειωθεί η πολιτική του δύναμη αυτή η ενέργεια του τούρκου δικτάτορα είναι οπωσδήποτε αντιδημοκρατική και πρόκειται να πυροδοτήσει νέα βία ήδη τεταμένη πολιτική κατάσταση της χώρας. Το ερώτημα το οποίο τίθεται όμως είναι γιατί ορισμένοι από εσάς εκπλήσονται και φαίνονται αγανακτισμένοι για αυτή τη συμπεριφορά του Προέδρου Ερντογάν. Εσείς δεν είσαστε αυτοί οι οποίοι μέχρι τώρα τον ανεχόσαστε να σας εκβιάζει και να σας απειλεί. Εσείς δεν τον εκλυπαρείτε ακόμη και τώρα για να συνεργαστεί μαζί σας ωστόσο ώστε να επιληθεί δεν θα το μεταναστευτικό. Εσεί δεν είστε αυτοί οι οποίοι ανέχθηκαν την ελληνική κυβέρνηση Σαμαρά να κάνει ακριβώ το ίδιο πράγμα το οποίο έκανε ο πρόεδρο Ερντογάν. Να κλείσει δηλαδή τον αρχηγό και του βουλευτέ, του τρίτου πολιτικού Κόμματο Χρυσή Αυγή στη φυλακή. Εσεί δεν είστε αυτοί οι οποίοι ακόμη και τώρα τον ανέχεστε να σα περιπέζει και να περιπέζει παράλληλα και την Ευρώπη. Ήθελα να ρωτήσω εάν σας απίφθινε αυτή την ερώτηση ο κύριος Ορντογάν, τι θα το απαντούσατε. και τέλος για να δούμε και σοβαρά το θέμα είστε αποφασισμένοι έχετε την αξιοπρέπεια να απειλήσετε την τουρκία ότι θα διακοπούν οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις της. έχετε την δυνατότητα να απειλήσετε την τουρκία ότι θα αφαιρέσετε το πκκ από τις τρομοκρατικές οργανώσεις. Κυρίες και κύριοι, η Ευρώπη χρειάζεται την Τουρκία και η Τουρκία χρειάζεται την Ευρώπη. Και βεβαίως και οι δύο πλευρές πρέπει να σέβονται τους κανόνες του παιχνιδιού, πράγμα το οποίο προς το παρόν δεν συμβαίνει η τροποποίηση του συντάγματος Τουρκίας ε, ώστε να στερηθούν την ασυλία ένα, ένα μεγάλο μέρος της ε, αντιπολίτευσης είναι έχει κίνητρα τα οποία θα έχουν και σοβαρές επιπτώσεις στο μέλλον. Ένας, ε, μια προϋπόθεση για να δοθεί στην Τουρκία η θεώρηση είναι η σωστή νομοθεσία διότι υπό... με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούσε να διωχθεί η νόμιμα εκλεγμένη αντιπολίτευση. Χθες είδαμε στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης ε, ε, ένα αποτέλεσμα της συμπεριφοράς της, της κυβέρνησης που είναι κατά της ε, οικονομικής πολιτικής. Η κυρία 1,5 λεπτό. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συζήτηση γίνεται μόνο μία μέρα μετά την τελευταία τρομερή τρομοκρατική επίθεση στην Κωνσταντινούπολη, οπότε θέλω να αναφερθώ στα θύματα, να έχουμε συνέστηση ότι η Τουρκία έχει ένα σοβαρό πρόβλημα τρομοκρατίας. Και η καταπολέμηση τρομοκρατίας πρέπει να συνεχιστεί, αλλά ποτέ δεν πρέπει να γίνει εις βάρος της δημοκρατίας και της ελευθερίας. Και αυτό είναι το μήνυμα κάθε στήριξη στην καταπολέμηση της, δημοκρα... τρομοκρατίας αλλά με σεβασμό της δημοκρατίας γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε ακούσει πολύ άσχημα πράγματα οι αυταρχικές τάσεις του Ερντοάν ε, επιβεβαιώνονται, διώκονται δημοσιογράφοι, νομικοί βέβαια η στάση του έναντι όλων των γυναικών της Τουρκίας είναι ιδιαίτερα υποτιμητική. Μόλις χθες ο κύριος Ερντογάν έκανε τέτοιες δηλώσεις και η άρση της ασυλίας πρέπει να είναι λόγος σοβαρής ανησυχίας, ανησυχίας διότι επιδεινώνεται η κατάσταση του κράτους δικαίου στην Τουρκία. Ο Ερντογάν θα πρέπει να σταθεί μια στιγμή, να επανέλθει στην οδό του διαλόγου, της δημοκρατίας και της προσπάθειας εξέβρεσης ειρηνικής λύσης. Και αν ε, ακολουθήσει αυτή την οδό θα μας βρει στο πλευρό του. Όσο δεν το κάνει δεν θα είμαστε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Χάνκελ ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε από τις περίπου 60 μουσουλμανικές χώρες η Τουρκία ήταν μία από τις λίγες που μέχρι πριν από λίγο ήταν, προς την, ήταν στην οδό προς τη δημοκρατία τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ισότητα ανδρών και γυναικών όμως ε, μόνο η Τινησία έχει απομείνει τώρα πλέον όπως κάθε δικτάτορ και ο Ερντογάν χρειάζεται αντιπάλους και τώρα είναι οι Κούρδοι το κόμμα του, το ΧΑΝΤΕΠΕ θα έπρεπε με πολύ σαφέστερο τρόπο να διαχωρίσει τη θέση του από την τρομοκρατική οργάνωση ΠΚΚ. Το ΧΑΝΤΕΠΕ ποτέ δεν θα έπρεπε να έχει συμμετάσχει ε, στην κηδεία ενός ε, τρομοκράτη που έκανε επίθεση αυτοκτονίας και που ήταν του ΠΚΚ όπου δολοφονήθηκαν Τούρκοι. Γιατί αλλιώ ε, διευκολύνει την κατάσταση ο Ντεμιρτά για τον Ερντοάν του επιτρέπει να του αντιμετωπίζει, να του παρουσιάζει ω τρομοκράτε και να επιβάλλει δικτατορία όχι μόνο επί των Κούρδων αλλά και επί όλων των Τούρκων. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Χρυσόγονο, ένα λεπτό. Το ημιαυταρχικό καθεστώ τη Τουρκία απομακρύνεται από τον κοινοβουλευτισμό και μεταλλάσσεται σε απροκάλυπτη δικτατορία. Ο κύριος Ερντογάν μαζί με τους υποτακτικούς του καλλιεργεί και εμπορεύεται συστηματικά το μίσος προκειμένου να παγιώσει την ομή της εξουσίας. διοργανώνει γιορτές μίσους στα βυζαντινά τείχη της κωνσταντινούπολης για να πανηγυρίσει την άλωσή της πριν από έξι περίπου αιώνες και τις σφαγές και λαιλασίες που επακολούθησαν. αρνείται να αποδοκιμάσει το μίσος των οθωμανών κατά των αρμενίων και των άλλων χριστιανικών πληθυσμών και να αναγνωρίσει τις γενοκτονίες που διαπράχθηκαν σε βάρος τους πριν από έναν αιώνα. διεξάγει και σήμερα έναν ακήρυκτο πόλεμο κατά της κουρδικής μειονότητας στις νοτιοανατολικές επαρχίες και αναιρεί την ασυλία των βουλευτών του κουρδικού κόμματος χαντεπέ με σκοπό να φημώσει γενικότερα την αντιπολίτευση. η ευρωπαϊκή ένωση πρέπει να μιλήσει στον κύριο ερντογάν στη μόνη γλώσσα που θα καταλάβει τη γλώσσα των πολιτικών και οικονομικών κυρώσεων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, Επίτροπε. 7η Ιουνίου είναι η επέτειος κατά την οποία πέρυσι οι πολλοί Κούρδοι βουλευτές μπήκαν στην ε, τουρκική εθνοσυνέλευση και αυτό γιατί τους ψήφισαν Κούρδοι αλλά και πολλοί άλλοι που ήθελαν να αλλάξει η κατάσταση. Δεν είναι λοιπόν σύμπτωση που χτες πέρασε ο νόμος που στρέφεται κατά των 138 βουλευτών των οποίων ήρθε η ασυλία με τόσο αντιδημοκρατικό τρόπο. Μοιάζει σαν, σαν εκδίκηση του Ερντογάν μετά την περσινή νίκη και αυτό είναι χτύπημα στο κράτος δικαίου της Τουρκίας. Θέλω λοιπόν η Επιτροπή να φροντίσει να μην επιτραπεί στην Τουρκία να ξεπεράσει αυτό το θέμα εν ώψη της απελευθέρωσης των θεωρήσεων. Δεν μπορούμε να στηριζόμαστε στην Τουρκία για την επίλυση προβλημάτων που έχουμε με τους πρόσφυγες και το θέμα της ελληνικής. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριο Κεφαλογιάννη για ένα λεπτό να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια και την έντονη ανησυχία για τις τελευταίες τρομοκρατικές επιθέσεις στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Θέλω επίσης να εκφράσω την έντονη ανησυχία αλλά και τη δυσφορία μου γιατί η τουρκική κυβέρνηση για πρώτη φορά μετά από 82 χρόνια, από το 1934, επιτρέπει την ανάγνωση του Κορανίου στη διάρκεια του Ραμαζανίου ε, μέσα στην Αγία Σοφιά αγιά σοφία η οποία είναι μνημείο της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και προστατεύεται από την unesco. θέλουμε μια τουρκία δημοκρατική θέλουμε μια τουρκία σταθεροποιητικό παράγοντα στην ευρύτερη περιοχή θέλουμε μια τουρκία η οποία να προσφέρει ασφάλεια και ευημερία στο λαό της. όμως η τουρκία είναι μια χώρα η οποία απομακρύνεται από τη δημοκρατία διολυσταίνει σε αυταρχικό καθεστώς με ισλαμικά στοιχεία είναι μια χώρα που δυστυχώς απομακρύνεται από την ευρωπαϊκή ένωση με ευθύνη της ηγεσίας της. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Μπενιφέ έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η συνταγματική αυτή μεταρρύθμιση που πέρασε από το ΑΚΠ στην Μεγάλη Εθνοσυνέλευση της Τουρκίας για την άρση της βουλευτικής ασυλίας 138 βουλευτών είναι κάτι πάρα πολύ ανησυχητικό. Μην ξεχνάμε ότι ο Ερντογάν μίλησε για ιστορική στιγμή για τη χώρα. Βλέπουμε ξεκάθαρα το που μακρύνει όλο και περισσότερο Ερντογάν από τις αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξέρετε ότι πριν από μερικές εβδομάδες προσπαθήσαμε εγώ και πολλοί άλλοι συνάδελφοι να ε, σταματήσουμε την πράξη αυτή που έλεγε χώρα τελικά στην Τουρκική Βουλή. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι υπάρχουν πάρα πολλές μυστικές υπηρεσίες στην Τουρκία, οι οποίες εκμεταλλεύονται το καθεστώς τρομοκρατίας προκειμένου να κάνουν διάφορες έρευνες και προκειμένου να επισύρουν ευθύνε πάνω στην αντιπολίτευση για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στη χώρα. Δεν μπορούμε λοιπόν αυτή τη στιγμή να συνεχίζουμε εμεί τη συνεργασία με την Τουρκία στα διάφορα θέματα τα οποία έχουμε ανοίξει. Ο κύριος Τζαμπάσκη έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, για άλλη μια φορά βλέπουμε ότι η Τουρκία με επικεφαλή στον Ερντογάν αποδεικνύει ότι δεν σέβεται καθόλου τις δημοκρατικές αρχές δεν μπορεί λοιπόν να έχει θέση η χώρα αυτή στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν προχωρά σε μια απόφαση άρση τη βουλευτική ασυλία 138 βουλευτών. Πραγματικό πλήγμα κατά τη δημοκρατία. Πρόκειται για μια πραγματική απόπειρα να στραφεί τελικά εντελώς κατά και να καταργήσει το φιλοκουρδικό κόμμα ΧΑΝΤΕΠΕ. Δεν θα μου κάνει εντύπωση αν όλα αυτά τελικά οδηγήσουν σε εμφύλιο πόλεμο στην Τουρκία μετά από όλες αυτές τις διαφορετικές επιθέσεις που έχουν λάβει η χώρα. Νομίζω ότι θα πρέπει πάση θυσία να σταματήσουμε την Ερντογάν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τη ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να παγώσουν κάθε διαπραγμάτευση με την Τουρκία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προασπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι λοιπόν τώρα η κατάλληλη στιγμή να αναλάβουμε δράση και να δείξουμε ότι η Τουρκία ως έχει αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να είναι τέρος μας. Αρίστη δεν είναι μόνο επίθεση κατά 138 βουλευτών όπως ήδη υπόθηκε, είναι μια απευθείας επίθεση κατά ε, των λίγων στοιχείων του δημοκρατικού πολιτεύματος που έχουν ε, απομείνει στην Τουρκία. Το είπε σαφώς η Γκάμπι Τσίμε. Ο Ερντοάν καταπατά κάθε δημοκρατικό δικαίωμα. Το σώμα θα πρέπει να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα όχι μόνο κατά τη ε, στρατηγική του Ερντοάν αλλά και υπέρ αυτών των βουλευτών. Υπέρ των πολιτικών δυνάμεων που απεγνωσμένα προσπαθούν να ξεκινήσουν ένα δημοκρατικό διάλογο σε αυτή τη χώρα. Είναι θεμελιώδες αυτό το τελευταίο στοιχείο, διότι ο Ερντοάν και ο στρατός καταπνίγουν και φημώνουν κάθε τέτοια δυνατότητα με αυτό το τελευταίο διοικητικό πραξικόπημα που έκαναν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανησυχεί ιδιαίτερα, αλλά πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα. Η συμφωνία με την Τουρκία σημαίνει ότι τα κράτη-μέλη δίνουν λεφτάρα και νομιμοποίηση στον Ερντοάν. Αλλά δεν λένε τίποτα για την άθλια κατάσταση των ε, προσφύγων που είναι παγιδευμένοι στην Τουρκία και για την ε, γενοκτονία των, και για τους ε, σφαγές των Κούρδων. Ο κύριος Κάρας, κύριε Επίτροπε. Όσο και αν δεν είμαι πεισμένο για τη συμφωνία αυτή Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για του πρόσφυγε, οι εξελίξει είναι ιδιαίτερα λυπηρέ, απαράδεκτε. Και αυτά που λέει το σώμα είναι απαραίτητα και σωστά. Όταν 138 βουλευτέ με μία ενέργεια νόμιμα εκλεγμένοι εκπρόσωποι της ε, αντιπολίτευσης βλέπουν την ε, ασυλία τους να έρεται όταν ε, μια πολιτική δύναμη της αντιπολίτευσης αποκλείεται από τη Βουλή όταν δεν μπορούν να ασκήσουν τα καθήκοντά τους όταν οι δυνάμεις αντιπολίτευσης κατηγορούνται για την πολιτική τους δραστηριότητα και σε μεγάλο βαθμό φημώνονται τότε δεν μπορούμε να πούμε ότι συνάδει αυτό με τις αξίες μας, ε, με το κράτος δικαίου. Οπότε πρέπει να το πούμε ανοιχτά. Η Τουρκία από πλευράς δημοκρατίας και από πλευράς κράτους δικαίου τα πάει στραβά και δεν θα υπάρξει συγγνώμη γι' αυτό. Ένα λεπτό κυρία Γκόμες. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βλέπουμε αυτή τη στιγμή πώ έχει κατάσταση στην Τουρκία. Βλέπουμε επίση όλε αυτέ τι τρομοκρατικέ επιθέσει, όπω η χθεσινή στην Κωνσταντινούπολη. Την καταδικάζουμε προφανώ. Δυστυχώ όλα αυτά τα γεγονότα συνδέονται μεταξύ του. Ο Ερντογάν αποφάσισε να άρει τη βουλευτική ασυλία 138 βουλευτών. Αυτό είναι σαφή επίθεση κατά των βουλευτών του ΧΑΝΤΕΠΕ. Στρέφεται κατά τη κουρδική μειονότητα ο Ερντογάν με την πράξη του αυτή και η τουρκική κυβέρνηση και κυρίως Ερτογάν ουσιαστικά με έναν εντελώ πρόδειλο τρόπο στρέφονται κατά τον ίδιο των κριτηρίων τη Κοπενχάγη, εφόσον δεν σέβονται καν τα πολιτικά δικαιώματα των βουλευτών. Δεν μπορεί να δεχθεί ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Συμβούλιο τον εκβιασμό αυτό του Ερντογάν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να δεχθούμε το ότι η χώρα αυτή μπορεί να θεωρείται μια ασφαλής χώρα όταν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Πρέπει λοιπόν αυτή τη στιγμή να δούμε τι θα καταφέρουμε, πώς θα καταφέρουμε να θεραπεύσουμε την κατάσταση στην Τουρκία. Μίκελς παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστώ πολύ. Πώς αντιδρά η Ευρώπη και οι Ευρωβουλευτές από αυτήν την απόπειρα ακύρωση του ίδιου του Κοινοβουλίου. Ο Τούρκος δημοσιογράφος Ζαν Τίντερ περιγράφει τη χώρα του ως εξής. Στην Τουρκία μπορείς να δράσεις ελεύθερα. Αν είσαι τετεθειμένος να πληρώσεις το τίμημα. Συγκεκριμένα, για τους βουλευτές τώρα του ΧΑΝΤΕΠΕ, αξιοποιείται νόμος ε, κατά της τρομοκρατίας. Διώκονται επειδή έχουν συμμετάσχει, για παράδειγμα, σε ειρηνικές διαδηλώσεις ορισμένοι. Έχει παρέλθει η ώρα των δηλώσεων και των εκκλήσεων. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο πρέπει να δράσουν. Ας αρνηθούμε ως Κοινοβούλιο την έγκρισή μας στην ε, απελευθέρωση των θεωρήσεων. Αλλά επίσης και οι βουλευτές στην Τουρκία αυτοί που διώκονται χρειάζονται άμεση στήριξη. Στη Γερμανία έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια, οι βουλευτές στηρίζουν βουλευτές. Α κάνουμε κάτι το παρόμοιο και εμείς εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να στηρίξουμε την ελπίδα για δημοκρατία στην Τουρκία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Μαυρίδης ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, οι κανόνες δικαίου και της δημοκρατίας έχουν προκαιρού συντριβεί στην Τουρκία. Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι κάτι πολύ περισσότερο και κάτι πολύ χειρότερο. Είμαστε μάρτυρες μιας γενοκτονίας σιωπηλής που γίνεται στις κουρδικές επαρχίες με εκατοντάδες δολοφονίες και αθώα θύματα. τώρα ο Ερτογάν προχωρεί και άρει την ασυλία των βουλευτών που διαφωνούν μαζί του. πρώτος στόχος ο αποκεφαλισμός της ηγεσία του ΧΤΠ, του κόμματος που είναι η μοναδική συγκροτημένη αντιπολίτευση. απέναντι στη βία όμως και την επιθετικότητα του Ερτογάν η αντιπολίτευση ιδίως οι κούρδοι αντιδρούν με ειρηνικά και πολιτικά μέσα. για κάθε ένα βουλευτή που θα διώκεται κάποιοι από εδώ μέσα είμαστε αποφασισμένοι να παρέχουμε προσωπική αλληλεγγύη και στήριξη και επίσης στηρίζουμε την απόφαση του χατεπέ όπως να αρνηθεί να προσέλθει σε ανάκριση μετά τα διατάγματα του ερντογάν. Η κυρία Σακοράφα για ένα λεπτό. Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Επίτροπε, η σημερινή συζήτηση επιβεβαιώνει παλιότερες επισημάνσεις μου. Διαχρονικά ωρεοποιείται και παραβλέπεται όσα τραγικά συμβαίνουν στην Τουρκία στο όνομα εξυπηρέτηση οικονομικών συμφερόντων και μικροπολιτικών επιδιώξεων εσωτερικής κατανάλωσης και απόδειξη είναι η συμφωνία για το προσφυγικό που καταγγέλθηκε από τον ΟΗΕ. Η πολιτική χαϊδέματος προς τον Ερντογάν και την τουρκική πολιτική ελίτ του επέτρεψαν να δημιουργήσει ένα αντιδημοκρατικό πλέγμα διώξεων οποιοδήποτε διαφωνεί πολιτικών αντιπάλων, ακαδημαϊκών, δημοσιογράφων και άλλων. Η ποινικοποίηση του κουρδικού ζητήματο με την παραποποίηση σε δίκη Κούρδων βουλευτών είναι η φυσική εξέλιξη. Αυτή τη χώρα ονομάζεται ασφαλή και με την ηγεσία τη διαπραγματεύεστε συμφωνίε τη. Ασφαλώ και είμαστε υποχρεωμένοι να αντιταχθούμε στι διώξει των Κούρδων βουλευτών. Το γεγονό αυτό όμω δεν είναι μεμονωμένο, κύριε Επίτροπε είναι ενταγμένο σε ένα συνολικό σχεδιασμό του ερντογάν και φοβάμαι ότι σύντομα θα βρεθούμε μπροστά σε χειρότερε εξελίξει που θα επηρεάσουν και την ευρύτερη περιοχή. η αναθεώρηση τη πολιτική σα λοιπόν με την επιβολή ακόμα και κυρώσεων είναι επιτακτική ανάγκη. ευχαριστώ κύριε πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Πιερ Αντώνιο Παντσέρη για 1,5 λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μετά την άρση της ασυλίας των βουλευτών και αφού το συνταγματικό δικαστήριο απέρριψε την προσφυγή που έκανε το ΧΑΝΤΕΠΕ, ο στόχος είναι ξεκάθαρος αυτή τη στιγμή. Να περάσουν από δίκη οι 50 αυτοί βουλευτές του ΧΑΝΤΕΠΕ και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να δούμε ότι ο Ερντογάν θέλει να αλλάξει τη φύση και τη φυσιογνωμία του τουρκικού κοινοβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν απέναντι σε όλα αυτά θα πρέπει να βγει από τις αντιφάσεις στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή, στην περίεργη σχέση που έχει με την Τουρκία. Τουρκία. Πρέπει αυτή τη στιγμή να χρησιμοποιήσουμε όλη τη διαπραγματευτική μας ισχύ για να εμποδίσουμε τέτοιες εξελίξεις. Δεν μπορούμε στο όνομα της σταθεροποίησης να δίνουμε πόρους προκειμένου να σταματήσει με την αισθητική ροή από την Τουρκία προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη στιγμή που η Τουρκία δεν συμπεριφέρεται πλέον δημοκρατικά. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όσο οποιαδήποτε συμφωνία έχουμε πλέον με την Τουρκία υπάρχουν υπάρχουν συγκεκριμένε προποθέσει όσον αφορά τα δημοκρατικά δικαιώματα. Μόνο κατά αυτόν τον τρόπο μπορεί να διεξαχθεί ο διάλογο με την Τουρκία. Ο κ. Παπαδάκη, παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η απόφαση για άρση της βουλευτική ασυλίας αποτελεί ακόμη μία αντιδημοκρατική κίνηση που έχει αναφυσβήτητα απότερο στόχο να ενισχυθούν εξουσίες του Ερτογάν. Με τη νέα διάταξη τα μέλη του ΧΑΤΕΠΕ όχι απλά μπαίνουν στο στόχαστρο αλλά ουσιαστικά δρομολογείται η εξάλληψη του κόμματο από το κοινοβούλιο. δεν μπορούμε να αποστρέφουμε το βλέμμα μπροστά στι παραβιάσεις της ελευθερία της έκφραση στην τουρκία με το φόβο ότι θα τεθεί σε κίνδυνο η συμφωνία Ευρωπαϊκή Ένωση Τουρκία για του πρόσφυγε υπενθυμίζω ότι η βουλευτή του χδπ λέιλα ζανά που έλαβε το βραβείο ζαχάροφ είχε μείνει για δέκα χρόνια στη φυλακή μετά από άρση της ασυλίας της το 1994. Η άρση της ασυλίας αποτελεί κατάφορη παραβίαση των δικαιωμάτων των βουλευτών και θα χειροτερέψει την ήδη υπάρχουσα τεταμένη κατάσταση σε σχέση με τον κουρδικό δυστυχώς τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά κατά της ελευθερίας της έκφρασης του αποκλεισμού του δημοκρατικού διαλόγου της φήμωσης του τύπου της συνεχιζόμενης κατοχής της κύπρου δείχνουν ότι η τουρκία είναι μακριά από τις αρχές και αξίες της ευρωπαϊκής ένωσης στην οποία θέλει να ενταχθεί. Περνάμε τώρα Όλοι οι συνάδελφοι που έχουν πει να πάρουν το λόγο θα τον πάρουν. Ο κύριος Σόλτς πρώτος. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα μπορούσαμε εκτενέστατα να συζητάμε το ζήτημα αυτό. Στη χώρα μου υπάρχουν πολλοί βουλευτές που προσπαθούν να κρυφτούν πίσω από την ασυλία και αποποιούνται κάθε ευθύνη που έχουν για συγκεκριμένες πράξεις τους. Όσον αφορά όμως τώρα την απόφαση στην Τουρκία δεν μιλάμε μόνο για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για το ότι πλέον ξεκάθαρα είμαστε απέναντι σε ένα μέτρο το οποίο στρέφεται στοχευμένα μια συγκεκριμένη μειονότητα και ενό συγκεκριμένου πολιτικού κόμματο. Αν λοιπόν η τουρκική ηγεσία αναλαμβάνει δράση προκειμένου να θέσει εκτός νόμου ένα πολιτικό κόμμα, αυτό σαφώς αποτελεί πλήγμα κατά των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου. Για μα υποτίθεται ότι αυτά τα δύο είναι σημαντικότητε αρχέ, άρα πρέπει να υπάρχουν επιπτώσει. Μέσω τη απόφαση αυτή η Τουρκία απομακρύνει το όλο και περισσότερο από τον δρόμο που θα μπορούσε να την οδηγήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε την κατάσταση και να αποσαφηνίσουμε ότι όντω η Τουρκία θα πρέπει να τηρεί τα δικαιώματα τη κουρδική μειονότητα. Άλλη εναλλακτική δεν υπάρχει. Όσον αφορά τώρα τι τάσει Ευρώπη, ε, λοιπόν, δεν μπορούμε να κάνουμε να μην συμβαίνει τίποτα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Καπούτο έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Με την άρση της βουλευτικής ασυλίας στην Τουρκία, πάνω από 100 βουλευτές της αντιπολίτευσης κινδυνεύουν να συλληφθούν. Βλέπετε αυτή τη στιγμή λοιπόν ότι η Τουρκία κατευθύνεται σε ένα αυταρχικό δρόμο και όλο και περισσότερο δεν νομίζουμε ότι το σύστημα, ακόμα και το δικαστικό, είναι αμερόληπτο και τετκειμενικό. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε λοιπόν ότι δεν τηρείται το κράτος δικαίου. Επίσης, πολύ περίεργη και επικίνδυνη σχέση της κυβέρνησης μαζί με τον, απέναντι στον τύπο και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι δέχονται όλο και περισσότερο, όχι μόνο απειλές, αλλά πολλές φορές ακόμα και σωματικές επιθέσεις. Απέναντι λοιπόν σε όλες αυτές τις πρόδειλες παραβιάσεις του κράτους δικαίου και των δικαιωμάτων, είναι πολύ σημαντικό να διαμορφώσουμε συγκεκριμένη στάση απέναντι στην Τουρκία και να δούμε τελικά αν και πώς η χώρα αυτή θα μπορούσε να πλησιάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση κυρία Κονέτσνα. Αγαπητοί συνάδελφοι, η Τουρκική Βουλή ενέκρινε μια συνταγματική μεταρρύθμιση για να άρει την ασυλία 138 βουλευτών. Ξέρουμε ποιους στοχεύουν αυτά τα μέτρα. Την αντιπολίτευση. Αλλά το θέμα είναι εάν ε, θα πρέπει να συνεχίσουμε την προσπάθεια φιλελευθεροποίησης των θεωρήσεων προς μια τέτοια χώρα που θίγει θεμελιώδη δικαιώματα, θίγει τα δικαιώματα όλων των πολιτών της και δηλαδή των Κούρδων και το οποίο κράτος ε, θέλει να ε, καταπνίξει κάθε φωνή στο, στην περιοχή των Κούρδων. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι λάθος να παραμένουμε σιωπηλοί και θέλω να μου πείτε λοιπόν τι θα κάνετε. Θα συνεχίσετε να κάνετε σαν να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αν το κάνετε αυτό θα επιδεινωθεί ακόμη περισσότερο η κατάσταση. Ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος. Ο κύριος Κόουσον. Περμούι. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ο Επίτροπος λέει ότι η Επιτροπή ανησυχεί. Τι πάει να πει ανησυχεί στην Άγκυρα δεν μοιάζει να ανησυχεί κανείς για την ανησυχία της ε, Κομισιόν. Γιατί έχετε κάνει συμφωνία για να υπάρξουν ε, τοπικές απελάσεις ε, προσφύγων. Οπότε δεν σα ενδιαφέρει τόσο πολύ το ότι έρεται η ασυλία του Χαντεπέ και άλλων τη αριστερά στην Τουρκία. Δεν κάνετε τίποτα από φασιστικό, το αποτελεσματικό κατά του κλεισίματο ΜΜΕ, τη σύλληψη δημοσιογράφων, των βομβαρδισμών αμάχων στι κουρδικέ περιοχέ και τη δράση γενικότερα του διαβόητου αντιτρομοκρατικού νόμου. Έχουμε λοιπόν αυτή την προσπάθεια ε, αποκλεισμού των ε, Κούρδων βουλευτών. Και εσείς τι κάνετε. Κάνετε άφλε συμφωνίες με τον Σουλτάν Ερντοάν. Και στην ουσία ε, δημιουργείται σε οποιαδήποτε προσπάθεια ειρήνευσης διατηρώντας το ΠΚΚ στην λίστα των, τρομοκρατικών οργανώσεων. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο Πρόεδρος. Κύριε Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίε και κύριοι. Η συζήτηση σαφώς κατέδειξε ότι υπάρχει κοινότητα απόψεων. Τουλάχιστον όσον αφορά το ότι είναι απαράδεκτη αυτή η απόφαση. Η απόφαση αυτή είναι αρθή ασυλία συλλογικά 138 βουλευτών. Εδώ δεν υπάρχει καμία παρανόηση. Είναι απαράδεκτο να γίνονται τέτοια πράγματα και δεν ανταποκρίνεται σε ένα κράτος δικαίου. Και εγώ ήμουν μέλο τη ε, Επιτροπή Άρση Ασυλία στο Εθνικό Κοινοβούλιο για πολλά χρόνια και ξέρω πέρα πρόκειται. Δεύτερον, κυρίε και κύριοι, είτε το θέλουμε είτε όχι, και πρέπει να το θέλουμε, πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι γεωγραφικά η Τουρκία είναι εκεί που είναι. Μετά την Ρωσία και μαζί με την Αίγυπτο, η Τουρκία είναι η πολυπληθέστερη χώρα στην άμεση γειτονία μας. 90 εκατομμύρια. Και έχει τη γεωγραφική θέση που έχει. Ως Ευρωπαϊκή Ένωση, ως υπεύθυνη για τη λήψη αποφάσεων στην Ένωση, πρέπει να συζητάμε με τους εταίρους μας, με τους γειτονές μας και να συζητάμε τα θέματα που πρέπει να συζητάμε. Για το θέμα των ε, ε, προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών χρειάστηκε να συζητήσουμε περισσότερο με την Τουρκία. Και υπάρχουν και άλλοι τομεί όπου πρέπει να υπάρξει περισσότερη συνεργασία με αυτήν την υποψήφια χώρα Τουρκία. Και από αυτήν την ε, ε αντίληψη προέκυψε το πρόγραμμα δράσης. Και το πρόγραμμα δράσης ε, περιέχει και την πλευρά πώς θα βοηθήσουμε την Τουρκία για να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση και νομίζω ότι πρόσφατα όλοι αναγνωρίζουμε ότι η χώρα φιλοξενεί πολλούς πρόσφυγες όπως και άλλες χώρες στην περιοχή και οι χώρες αυτές ε, πρέπει λοιπόν να λάβουν την αναγκαία στήριξη από μας. Επίσης το πρόγραμμα δράσης αναγνωρίζει ότι οι ενταξιακές διαπραγματεύσεις πρέπει να επιταχυνθούν να αποκτήσουν ε, νέα όθηση και γι' αυτό πρέπει να προχωρήσει και η φιλελευθερωποίηση των θεωρήσεων. Η Τουρκία ε, η ίδια έκανε αίτηση. Θέλει να γίνει μέλο τη Ένωση. Δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει μέλο τη Τουρκία. Και η Τουρκία θέλει φιλελευθερωποίηση των ε, ε, θεωρήσεων για τους Τούρκου πολίτε που θέλουν να ταξιδεύουν στην Ευρώπη. Αφόσον αυτή είναι η επιθυμία τη, τότε το συζητάμε. Αλλά θέτουμε και προποθέσει. Και αν οι προποθέσει δεν πληρούνται, τότε δεν προχωράει το θέμα. Έτσι γίνονται τα πράγματα αυτά το αντιμετωπίζω όπως και πολλοί από εσά η Τουρκία παρά το ότι πάντα εκφράζει την επιθυμία να γίνει μέλος της Ένωσης κινείται προς άλλη κατεύθυνση, εντελώς άλλη και θα ήθελα να μάθω να μας πει σαφώς ο κύριος Ορντοάν που είναι τόσο σημαντικός σε αυτή τη χώρα εάν εξακολουθεί να το θέλει ή όχι γιατί είναι κρίμα να χάνουμε το χρόνο μας εμείς είμαστε διατεθειμένοι αλλά μόνο με βάση τις προϋποθέσεις μας. Κράτος δικαίου, δεν είναι διαπραγματεύσουμε αυτό. Δεν υπάρχει τουρκική εκδοχή της δημοκρατίας. Υπάρχει μια ενιαία αντίληψη για τη δημοκρατία και τους κανόνες της. Όπως ε, το θεωρούμε εμείς στην Ευρώπη και στα κράτη-μέλη της Ένωσης. Όπως ακριβώς ασκούν τη δημοκρατία τα κράτη-μέλη της Ένωσης. Πρέπει νομίζω να έχουμε περισσότερη αυτοπεποίθηση. Κανένα ε, δεν πρέπει να φοβάται τον πρόεδρο Ντρογάν στην Ευρώπη, ούτε εγώ ούτε εσεί, Φαδίζουμε το δρόμο μα, έχουμε τι αρχέ μα, τι διαδικασίε μα. Μα ενδιαφέρει να έχουμε καλέ ε, σχέσει γειτονία, αλλά τότε πρέπει να γίνονται και οι αναγκαίε ενέργειε. Αυτές είναι οι πεπιθήσει, αυτέ είναι οι αρχέ τη Κομισιόν και να είστε βέβαιοι ότι σε καμία περίπτωση δεν θα αποχωρήσουμε σε κανένα από αυτά τα θέματα, αλλά επίση δείξτε κατανόηση διότι ε, εφόσον είναι γείτονά μα πρέπει να συζητάμε γιατί είναι και προς το συμφέρον σε τελευταία ανάλυση και των δικών μας συμπολιτών. Ευχαριστώ. Στο σημείο αυτό έληξε η συζήτηση και περνάμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι η δήλωση